δική του ενακτήρια του παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ. Όταν σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι προσέβλεπα να σας στην ε, επόμενη συνάντησή μας, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Στα αγγλικά πρέπει να προσέχει κανείς τι εύχεται γιατί μπορεί να του έρθει στο κεφάλι. Εδώ είμαι πάντως ενώπιόν σας. Χαίρομαι που έχω επιστρέψει ενώπιόν σας και είναι κατά κάποιο τρόπο μια προκαταβολή αυτών που ελπίζω να γίνουν στο μέλλον, δηλαδή μιας καρποφόρας και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ μας. Νομίζω ότι έχετε δει τις ε, απαντήσεις μου, τις λεπτομερείς απαντήσεις στα 23 πρόσθετα ερωτήματα που θέσατε. Καταρχήν όμως θα ήθελα να κάνω, αν μπορώ, ένα βήμα πίσω και να σας ζητήσω να φανταστείτε ότι είναι το 2019. Βρισκόμαστε ενώπιον των επομένων ευρωεκλογών και φτάνουμε στο τέλος της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ. Ή προς το τέλος της ε, θητείας της πρώτης Επιτροπής Γιούνκερ. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που μπορούμε να δώσουμε στους ψηφοφόρους μας. Τι πετύχαμε με τη συνεργασία μας για τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Η συνολική λοιπόν εικόνα για το 2019 θα είναι η Ευρώπη γύρισε στην ανάπτυξη. Μειώνεται η ανεργία, ιδίω η ανεργία των νέων. Οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που πέρασαν πολλές χώρες, ιδίως στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ευρώπης, οι κρίσεις αυτές έχουν περατωθεί, έχουν τελειώσει. Γυρίζουν οι χώρες αυτές σε οικονομική υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερη και πιο συνεκτική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και πολιτικές ανησυχίες των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά παραμένει μια οικογένεια 28 κρατών μελών μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εκ νέου επιτύχει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μια ισχυρή τραπεζική ένωση που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια ισχυρότερη και καλύτερα διαχειριζόμενη ζώνη του ευρώ και έχουν δώσει μεγαλύτερη ακτινοβολία στο ευρώ σαν παγκόσμιο νόμισμα. Με την υποστήριξη τη Κομισιόν, όλο και περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση. Η εμπιστοσύνη χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών που είναι μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην ε, ε, Τραπεζική Ένωση, μάλλον και αυτών που δεν είναι μέσα, επί τη βάση ενό κοινού ε, βιβλίου κανόνων για τα τραπεζικά θέματα. Καμιά τράπεζα δεν είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να επιτραπεί η αστοχία της έχουμε εξασφαλίσει την πολυμορφία του τραπεζικού συστήματος. Έχουμε και πάλι τράπεζες με ισχυρότερους ισολογισμούς και που δανείζουν στην υπόλοιπη οικονομία γιατί έχουμε εξασφαλίσει τις σωστές διαρθρωτικές αλλαγές. Οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζες και στην ασφάλεια των καταθέσεών τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζεται ως ένας ε, επόπτης παγκόσμιας εμβέλειας. Οι δοκιμασίες αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής την χάνουν εμπιστοσύνη και δίνουν μια σωστή ανάλυση τη υγεία των τραπεζών. Οι καταναλωτέ χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη επιλογή ασφαλέστερων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε χαμηλότερο κόστο όπω συντάξει και ασφαλίσει. 60 χρόνια μετά από την έγκριση τη συνθήκη τη Ρώμη, επιτέλου βλέπουμε την ανάδυση μια ενιαία αγορά κεφαλουχικών προϊόντων. Την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Έχουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που προστατεύει τους καταναλωτές και τους επενδυτές και δίνει εμπιστοσύνη και σωστό πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη, καλά διαχειριζόμενη, διάφανη και ρευστή αγορά κεφαλαίων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά η Ευρώπη χαίρεται και είναι υπερήφανη για το σύστημα χρηματοπιστωτικών της υπηρεσιών που εμποδίζει ανεύθυνη ανάληψη κινδύνου και βραχή ε, βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση, όπως έγινε στο παρελθόν, αλλά επιτρέψει στις εταιρείε να, να καινοτομούν και να επενδύουν με σόφρονα τρόπο μακροπρόθεσμα. Επίσης χαιρόμαστε για το ρόλο μας στη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός στεναρού συνόλου διεθνών κανόνων για τις χρηματαγορές που αναγνωρίζονται από όλους και ιδίως στις ταχαίως αναδυόμενες οικονομίες. Πάνω απ' όλα, το 2019 θα είμαστε υπερήφανοι για το ρόλο μας στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επί τη βάση της αξίας τους και όχι επί τη βάση της χώρας στην οποία λειτουργούν. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι αυτέ που δημιουργούν τι περισσότερε θέσει απασχόληση, αντιμετωπίζουν τι μεγάλε εταιρείε και με το να διαμφισβητούν το status quo κάνουν την οικονομία μα και την κοινωνία μα πιο ασφαλή και είναι οι πολίτες οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα κερδίσουν περισσότερο από την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξαναγυρίζω όμως το 2014. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι δεν θα υπάρξουν δυσκολίες στον δρόμο μπροστά μας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν ε, απόψεις για τις οποίες είναι απόλυτα πεπισμένοι και επιχειρηματολογούν υπέρ αυτών. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, γιατί πολλά από τα δομικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για το μέλλον αυτό υπάρχουν ήδη. Αν συνεργαστούμε και παραμείνουμε πιστοί στην πορεία μας, πιστεύω μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική, σταθερή και παγκόσμια ανταγωνιστική ε, ε, περιοχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ένα κλάδο ο οποίος θα μπορεί να χρηματοδοτεί τη μακροχρόνια ανάπτυξη και δίνει περισσότερα ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή αυτή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για τη μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε μια μεγάλη συνεισφορά στην Ευρωζώνη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Πράγματι όλα αυτά θα απαιτήσουν σημαντική κοινή εργασία. Γνωρίζω όμως ότι η Επιτροπή σας είναι συνηθισμένη σε αυτή τη συνεργασία. Θέλω να, να συνεχίσω το έργο του Μισελ Μπαρνιέ, να δημιουργήσω ε, εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και φυσικά και με τα κράτη-μέλη. Εάν με εγκρίνετε στο αξίωμα αυτό από την 1η Νοεμβρίου, έχω να σας δώσω μια απλή υπόσχεση. Θα είμαι ένας Ευρωπαίος Επίτροπος και για όλες τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεργαστώ μαζί σας όσο μπορώ πιο σκληρά και όπως ξέρω να εργάζομαι για να μπορέσω να κάνω αυτό το όραμα πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.